Καλησπέρα σας. Το επόμενο θέμα είναι η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και όπως ε, και στο παρελθόν καλώ τους ε, ευρωβουλευτές οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν να μπορέσουν να έρθουν μπροστά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάθονται υποχρεωτικά στη θέση τους. Εάν έρθουν πιο μπροστά ίσως ε, έχουμε μια πιο ζωντανή ανταλλαγή απόψεων. Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν ρωτάτε επιπρόσθετες ερωτήσεις έχετε μόνο 30 ε, δευτερόλεπτα για να δευτερολογήσετε. Καταρχήν θα μιλήσουμε για την ευημερία των ζώων και δίνω το λόγο στην κυρία Μάλστρεμ για να απαντήσει στο πρώτο ερώτημα και την ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόκειται να απαντήσω στην ερώτηση της Μαρίαν Χάρκιν. Συμφωνούμε με την ανησυχία ε, που έχει σχετικά με την ευημερία των ζώων ε, και έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα για ευημερία των ζώων μέσα στην κοινωτική νομοθεσία με τέτοιες δράσεις. Συνεχίζεται η συζήτηση δε στο Συμβουλίο για αυτό το θέμα και και στον τομέα της γεωργίας ε, συνιστά προτεραιότητα το θέμα για μας. Ε, θα υπάρξει και ειδική διάσκεψη για την ευημερία των ζώων στην Ουψάλα στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Ε, εκεί θα συζητηθούν τα τελικά πορίσματα του Welfare Quality, ενός προγράμματος που ζητήθηκε από την κοινότητα ε, για να εκπονηθεί ένα ε, σύστημα που θα αξιολογεί κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη η ευημερία των ζώων ε, στον τομέα της γεωργίας. Αυτό φυσικά θα είναι ευνοϊκό όχι μόνο στον τομέα της γεωργίας αλλά γενικότερα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 40 πανεπιστημιακά ιδρύματα από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Επίση, στη διάσκεψη θα συζητήσουμε το πόσο μπορούμε παγκοσμίω να αναβαθμίσουμε την ευημερία των ζώων. Μιλάμε για διεθνή διεθνείς οργανώσεις όπως ο ΦΑΟ, ο ΠΟΕ, ε, η διεθνή βιομηχανία, ε, ο κρέατος ε, και των προϊόντων κρέατος και ούτω καθεξής. Ε, και επίσης για, ε, μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Συμβούλιο πρόκειται να εγκρίνει σχετικά συμπεράσματα. Επίσης θα γνωρίζετε ότι θα πρέπει να υποβληθεί νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς προς το παρόν ε, επεξεργαζόμαστε την πρόταση για μια νέα οδηγία για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς λόγους δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που πρόκειται να επεξεργαστεί το Σύμβουλο κατά τη διάρκεια τη Σουηδική Προεδρία. Σα ευχαριστούμε, κυρία Χάρκιν. Επερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, καλησπέρα κυρία Μάλστρεμ. Χαίρομαι ότι λέτε ότι θέλετε να, να συνεχίσει η συζήτηση γιατί ουσιαστικά η νομοθεσία η οποία υπάρχει ισχύει μόνο από δύο ετών και στην Ιρλανδία δεν έχουμε ακόμη ετοιμαστεί, δεν έχουμε συστήματα μεταφορές, ε, έχουμε λήψεις και ε, εάν ε, προχωρήσουμε θα υπάρξει ανταγωνισμός οπότε ε, είναι λογικό να αλλάξουμε νομοθεσία η οποία ισχύει μόνο από δύο ετών ε, θα χρειαστούν όμως πρώτα επιστημονικά στοιχεία να αποδείξουν ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν, Υπουργός. Όπως είπατε είναι βασικό να αξιολογήσουμε σωστά όλα αυτά, να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα, διότι μέχρι τώρα ε, συγκεντρώνουμε επιστημονικές πληροφορίες και στην Ουψάλα έχουμε καλές επιστήμονες ε, για να συζητήσουμε ε, στο συνέδριο το θέμα αυτό και να αποτελέσει τη βάση για την απάντηση την οποία θα δώσει το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά χαιρετίζω και τις απόψεις του Κοινοβουλίου από αυτού, διότι θα είναι ένα καλό σημείο ενάρξεως μιας ε, κουβέντας. Έχω και δύο επιπρόσθετες, θα τις πάρουμε μία μετά την άλλη από την κυρία Μαγκίνες και τον κύριο Κάλλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ένα θέμα. Ελπίζω ότι η επιστήμη θα υπερισχύσει των αισθημάτων στη μεταφορά των ζώων και θα παρακαλούσα να ασχοληθείτε με την μεταφορά των αλόγων που δεν έχει εξεταστεί επαρκώς και μας απασχολεί τώρα και πιστεύω ότι η ευμερία των ζώων εις τα αγροκτήματα ίσως ε, ε, θα μπορέσει να βελτιωθεί ε, για τις τεράστιες επιδοτήσεις τις οποίες λαμβάνουν οι αγροκτήμονες οι οποίοι βοηθούνται χωρίς να έχουν ένα εισόδημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλλο. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό είναι αμφιλεγόμενο στην Ιρλανδία, ιδίω ε, ε, για αυτού οι οποίοι είναι υπέρ τη καταψηφίσεω της δίκη της Λισαβόνα και ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε χαμηλές τιμές ε, για το βοδινό κρέας. Μπορείτε να μας πείτε αν ε, θα υπάρξει κάποια λύση πριν από τις 2 Οκτωβρίου που θα ψηφιστεί το δημοψήφισμα για την Ιρλανδία. Αντιλαμβάνουμε τις απόψεις σας και τους πολίτες αλλά δεν μπορώ να σας ε, ε, υποσχεθώ ότι όλα αυτά θα λυθούν πριν από το δημοψήφισμα περιμένουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόλις ε, μας υποβληθεί θα ξεκινήσει η συζήτηση περιμένουμε όμως ακόμη την πρόταση αυτή και όλα αυτά τα κάνουμε ψυχρό δηλαδή χωρίς συναισθηματισμούς για να δούμε πώς καλύτερα μπορεί να λυθεί το πρόβλημα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Τώρα προχωρούμε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο είχε τεθεί αρχικώς από τον κύριο Μωράης και τώρα έχει αναλυφθεί από τον κύριο Χέτ σχετικά με την εμπορία των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κύριε Υπουργός, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Σουηδική Προεδρία συμμερίζεται την ανησυχία του κ. Μουράσα για την εμπορία παιδιών, για την σεξουαλική του εκμετάλλευση ή για άλλου στόχου. Είναι η σύγχρονη σκλαβιά. Εξαιρετικά επικερδή δραστηριότητα τη οργανωμένη εγκληματικότητα. Δηλώνουμε αποτροπιασμό όταν συμβαίνει αυτό είτε στην Ένωση είτε στον κόσμο. Η εμπορία, η σώματα εμπορία είναι, ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή ηταν ανεκαθεν ενα σημαντικο ζητημα στην ευρωπαικη ενωση και πρέπει να συνδυάσουμε δώσουμε διάφορα μέτρα για να καταπολεμήσουμε την παραβίαση των βασικότερων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, θα πρέπει να αναλάβουμε προληπτικά μέτρα, να καταπολεμήσουμε την οργανωμένη εγκληματικότητα και να προστατεύσουμε και τα θύματα. Η κοινοτική διέσμευση ε, σε σχέση με την καταπολέμηση της σωματεμπορίας ε, σχετίζεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και τη χρήση μη δεσμευτικών εργαλείων. Το 97 παραδείγματος χάρη κοινό μέτρο για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Ε, έχουμε την απόφαση πλαίσιο του 2002 επίσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Υπευλήθη δε νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη και την καταπολέμηση της και την προστασία των θυμάτων. Και έτσι θα καταργηθεί και η απόφαση πλαίσιο του 2002. Ο στόχο ε, είναι να ε, ε, προστατεύσουμε τα ευπαθή θύματα, κυρίω τα παιδιά και να βελτιώσουμε τις διατάξεις του ποινικού δικαίου για να ελαχιστοποιήσουμε την δευτερογενή θυματοποίηση. Ε, δηλαδή καλύπτονται όλους ιδιαίτερως ε, πλέον μέσα σε αυτή την πρόταση ανάγκες ε, των παιδιών. Επίσης έχουμε την απόφαση πλαίσιο για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, την παιδική πορνογραφία και ο στόχος είναι να έχουμε ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και ε, να επιβάλλουμε ισχυρότερες ε, κυρώσεις για τους ε, αυτούργους, για τους δράστες. Υπάρχει το πρωτοκόλλο του Παλέρμου επίσης και η σύμβαση, η σχετική σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και διάφορα άλλα διεθνή νομικά εργαλεία σε συνεργασία με την Υπουργική ειδική διάσκεψη που διοργανώσαμε ε, που, για τον Οκτώβρη για το θέμα αυτό. Έχουμε και την έκθεση από τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωματών που θα εκπονήσει μια έκθεση και θα συζητηθεί και θα προκύψουν συμπεράσματα ε, του Συμβουλίου για το θέμα της ε, ε, ε, σώματεμπορίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Στοχόλμης και θα συζητηθούν από το Συμβούλιο συνολικά το Δεκέμβριο. Ευχαριστούμε. Κύριε Χέρντα, ευχαριστώ Υπουργέ. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα και στην ε, Σουηδία, αλλά όχι μόνο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τη συζήτηση αυτού του ζητήματος τα τελευταία χρόνια. Θα θέλαμε απλά να τονίσουμε ότι είναι κρίμα ότι θα γίνει αυτή η διάσκεψη 19 και 20 Οκτωβρίου και εμείς εδώ οι ευρωβουλευτές δεν μπορούμε να είμαστε εκεί γιατί ε, ε, θα γίνει η σύνοδος τότε και δεν μπορούμε να παρευρεθούμε, αλλά τι να κάνουμε. Επίσης ξέρω ότι η Σουηδική Προεδρία είπε ότι θέλει να συζητηθεί το θέμα της εκμετάλλευσης των παιδιών σε σχέση με τον τουρισμό ε, και αυτό θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, δηλαδή θα υπάρξει η μόνιμη διεθνή σε ομάδα που θα συνεδριάσει εκείνη την ημερομηνία αλλά ε, ακριβώς γιατί θα κάνετε εσείς την παρέμβαση ε, σε αυτή τη συνεδρία. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ την Άννα Ξέρω πόσο αφοσιωμένη είναι σε αυτό το τομέα. Ε, είναι ατυχές ε, που συμπίπτει η διάσκεψη στη Σουηδία με την Σύνοδο της Ολομέλειας. Αλλά είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Γι' αυτό τη διοργανώνουμε τότε τη διάσκεψη. Λυπούμεθα για το δεύτερο ερώτημά σας, συγγνώμη δεν είμαι ενημερωμένη, θα το ελέγξω και θα σας απαντήσω γραπτός. Ευχαριστώ. Thank you. I have uh, further... Ευχαριστώ. Κυρία Λίμ, η κυρία Λίμ παρακαλώ. Ευχαριστώ για την απάντηση και εμένα με λυπεί το γεγονός ότι δεν μπορούμε να παραστούμε στη διάσκεψη αυτή γιατί είμαστε εδώ αλλά θα μπορούσατε να διασφαλίσετε στην ημερήσια διάταξη να συμπεριληφθεί η να τονιστεί ιδιαίτερα η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να διασφαλίσουμε μια ορατή ε, και ε, επίκαιρη θέση στην μυρίσια διάταξη αυτού του θέματος. Ευχαριστώ ναι, κυρία Λίν, θα το θέσω υπόψη των ε, οργανών της ε, διασκέψεως. Ευχαριστώ. Καλώς. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Κυρία Μαγκίνες, μήνυμα για την συνεδρίαση υψηλού επίπεδου της ΦΑΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, η διάσκεψη της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ΦΑΟ θα συνεδριάσει 18 Νοεμβρίου και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τη ημερήσιας είναι μεταρρύθμιση του οργανισμού που βασίζεται σε ένα ε, πρόγραμμα μέτρων ε, που εγκρίθηκαν το 2008 από όλα τα κράτη-μέλη του ΦΑΟ. Αυτό το σχέδιο δράση ε, συνεπάγεται μεταρρύθμιση με πολλού και διαφορετικού τρόπου. Μεταξύ άλλων, οι μελλοντικέ δραστηριότητε του ΦΑΟ θα καθοδηγούνται από τα αποτελέσματα τη αξιολόγηση του διαχειριστικού συστήματο με στόχο την αύξηση τη αποτελεσματικότητα ε, και την καλύτερη αξιοποίηση των φυστάμενων πόρων. Επίση, τα μεταρρυθμιστική διαδικασία θα έχει μακρόπνοε επιπτώσει στι δραστηριότητε ε, του ΦΑΟ σε σχέση με του ανθρώπινου πόρου και την αποκέντρωση των διαδικασιών του. Ε, κάποια ε, ζητήματα σχετίζονται με την τροποποίηση του κανονισμού ε, του ΦΑΟ σε σχέση επίσης υπάρχουν άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την επισητιστική ασφάλεια και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία παγκόσμιας ε, εταιρική σχέσης ε, για την επισητιστική ασφάλεια. Για να συζητηθούν αυτά τα θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο διοργανώνεται ε, η διάσκεψη στη Ρώμη στις 16 με 18 Νοεμβρίου από το ΦΑΟ. Εκεί θα κάνει δήλωση η Προεδρία μας. Ε, θα βασιστούμε στα ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου που υπάρχουν για την επιστημιστική ασφάλεια. Στις 11 Νοεμβρίου του 2008 αναγνώρισε το Συμβούλιο ότι η τωρινή διατροφική κρίση συνεπαγείται ότι είναι αναγκαία η συντονισμένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεργασία ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα ε, και μην ξεχνάτε και το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπλήρωση των στόχων τη χιλιετία ε, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008. Καλωσορίζουμε μέσα στα συμπεράσματα ε, την μεταρρυθμιστική διαδικασία του ΦΑΟ που προάγεται από όλα τα κράτη-μέλη του οργανισμού στα πλαίσια τη διαχειριστική επιτροπή του ΦΑΟ. Σε αυτή τη σύνοδο κορυφή υπάρχει ένα σαφή πολιτικό στόχο να βελτιωθεί το σύστημα που ακολουθεί ο ΦΑΟ για να κατοχυρωθεί η επιστημιστική ασφάλεια ε, και να αναλάβει το SFS ένα ηγετικό ρόλο. Η Προεδρία θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, στραφούμε προς το μέλλον για να διαχειριστούμε την τωρινή κρίση και για να εκπληρώσουμε ε, τον πρώτο στόχο της χιλιετίας, δηλαδή την κατάργηση της ένδυας. Ε, χρειάζεται μεγάλη αφοσίωση και δέσμευση από σε όλων. Η Προεδρία μας θεωρεί ότι η Σύνοδος Κορυφής ε, θα έπρεπε να έχει αυτό το σαφή πολιτικό στόχο, να υπάρχει ένα νέο σύστημα ε, για τον ε, εφοδιασμό με τρόφιμα των λαών όλου του κόσμου και θεωρούμε ότι στην Σύνοδο Κορυφής πρέπει να έχουμε να εγκριθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα για να καταπολεμήσουμε την τωρινή κρίση και να αυξηθούν οι παρεμβάσει, ώστε επιτέλου να εκπληρωθούν οι στόχοι τη χιλιετία. Ευχαριστούμε, κυρία Μαγκίνε. Αντιλαμβάνομαι και ευχαριστώ για τη λεπτομερή απάντηση, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η στάση της ε, Σουηδικής Προεδρίας για την κοινή γεωργική πολιτική επιμένοντας ε, να υπάρξει παγκόσμιος ε, επιστησική ασφάλεια. Είναι σκόπιμο να έχουμε μία τέτοια πολιτική στην Ευρώπη για να εξασφαλίσουμε την επιστημική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει σε αυτό το συνέδριο ή ε, το Συμβούλιο αλλά προφανώς η ΚΑΠ μπορεί ε, να βοηθήσει ιδίω στο μέλλον όταν θα την συζητήσουμε θα μπορέσει να διευκολύνει τις πιο ε, φτωχές χώρες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην κοινή αγορά και θα μπορέσουμε κατά τον ίδιο τρόπο να βοηθήσουμε ε, την εξάλληψη της ε, παρούσης ε, σαφούς κρίσεως και οξίας κρίσεως. Τώρα έχουμε διάφορες εκθέσεις από τις διάφορες χώρες και θα πρέπει να τα εξετάσουμε για να δούμε πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την μελλοντική κάπως τροποποιημένη κοινή γεωργική πολιτική για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν. Κυρία Υπουργέ, εδώ μιλάμε ε, για την επιστημιστική ασφάλεια αλλά εγώ θα ήθελα να αναφέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιστημιστική ασφάλεια που εξαρτάται από την παραγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σήμερα είχαμε μία συζήτηση με την κυρία Φίσερ Μπολ επί του θέματος και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013. Υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη. Ε, ίσως δεν έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε απόψε, αλλά είναι πολύ βασικό για τους γεωργούς. Κάπως απαντήσατε απαντήσατε στην ερώτηση, αλλά θα ήθελα να έχω από τους συναδέλφους σας περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, όντως είναι μια τεράστια συζήτηση και περίπλοκη αναφέρουμε στο συνέδριο ενώ εδώ μιλούμε για πιο γενικά θέματα. Δεν έχουμε ε, στόχο να ε, αποκρύψουμε κάτι αλλά περιμένουμε ορισμένα στοιχεία για το μελλοντικό προϋπολογισμό πράγμα το οποίο ε, περιμένουμε ακόμη όπως είχε συμφωνηθεί στο Συμβούλιο το 2004 περιμένουμε επίσης την ε, έκβαση και τον απολογισμό των δαπανών του προϋπολογισμού ιδίως αυτού του τεραστίου προϋπολογισμού και έχουμε καθυστερήσει ελπίζουμε ότι θα έχουμε τα στοιχεία πρώτου τέλους του έτους για να μπορέσει να γίνει η πρώτη συζήτηση μεταξύ κρατών μελών αλλά ουσιαστικά η Ισπανική Προεδρία είναι αυτή η οποία θα επεξεργαστεί τα κατά μέρους θέματα. Ευχαριστώ. Τα επιμέρους θέματα. Τώρα προχωράμε στην επόμενη ερώτηση της κυρίας Κράτσα, την οποία αντιπροσωπεύει απόψε η κυρία Γιαννάκου σχετικά με τη Συμφωνία Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Αυτό το θέμα το συζητήσαμε και νωρίτερα σήμερα. Δεδομένης της κρίσης, ε, οι αρχές έχουν αναλάβει έκτακτα μέτρα ε, για ε, να στηρίξουν τα δημοσιονομικά. Ήταν σωστά τα μέτρα και διαδραματίσαν σημαντικό ρόλο για να αποφύγουμε ακόμη σοβαρότερε κρίσει, να σταθεροποιήσουμε την οικονομία και να βελτιώσουμε τι οικονομικέ συγκυρίε. Αλλά η σταθεροποίηση τη χρηματοπιστωτική κατάσταση δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ύφαση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ούτω ώστε στο μέλλον να έχουμε την απαραίτητη υποστήριξη για την ανάκαμψη, ελπίζουμε να έρθει, ε, και να ε, στηρίξουμε την βιωσιμότητα, την μεσοπρόθεσμη και την βραχυπρόθεσμη των δημοσίων Σοσιοοικονομικών. Πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτούς τους δύο στόχους. Και γι' αυτό το 2005 επιτράπει αυτή η ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητα. Σε χαλεπού οικονομικού καιρού ε, ε, πρέπει να αναλυθούν τα απαραίτητα μέτρα για να τονώσουμε την οικονομική δραστηριότητα ε, και για να ξεκινήσει η ανάκαμψη θα πρέπει να έχουμε βιώσιμα δημόσια οικονομικά και να εξηγιάνουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς μας. Η κατάσταση διαφέρει πολύ από κράτο σε κράτο. Θα υπάρξουν διαφορετικά σχέδια, διαφορετικά χρονοδιάγραμμα ε, για να, ε, τον, για να βελτιώσουμε την οικονομική ε, πολιτική και να στηρίξουμε τα δημοσιοοικονομικά. Ε, υπάρχουν διάφορες συστάσεις που θα γίνουν σε επιμέρους ε, κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει μελλοντικά να, όλοι να σέβονται το υφιστάμενο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και εξού και η συζήτηση ε, το φθινόπωρο στο ΕΚΟΦΗΝ για τον απαιτούμενο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. και αναμένουμε αυτές οι συζητήσεις να οδηγήσουν σε σαφή ομοθυμία σχετικά με την εξυγίανση των ε, δημοσίων οικονομικών, ώστε να ε, έχουμε μακρόπνοη ε, αηφορία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ για τη σαφήνεια της απάντησής σας. Θα ήθελα να δώσετε μια ιδιαίτερη σημασία για το αν πρέπει να επιμείνουμε ώστε το 2010 να είναι έτος δημοσιονομικής εξυγίανσης ή να υπάρξουν κατά κάποιο τρόπο παρατάσεις ή καθυστερήσεις. Πράγμα που μέχρι σήμερα βέβαια στις πολιτικές δεν έχει ωφελήσει ιδιαίτερα την Ένωση Είναι δύσκολο, δύσκολο το ερώτημα αυτό. Ε, η διάσκεψη G20 θα συζητήσει τις exit strategies για να βγούμε από την κρίση. Έτσι θα αρχίσει η συζήτηση. Αλλά ξαναλέω, διαφέρει η κατάσταση από κράτος σε κράτος σε μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό θα έχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να εκινήσουμε τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι συνάρτηση ε, της ε, χρηματοοικονομικής ε, κατάστασης. Βλέπουμε το φως στην άκρη του τούνελ. Ε, έχουμε ελπίδα ε, και θέλουμε να κατευθυνθούμε προς αυτή την προσέγγιση του exit strategy. Και πρέπει να κινηθούμε ε, ταχύτατα γιατί οι πλέον άποροι θα πληγούν, θα έχουμε μεγάλο κίνδυνο ανεργίας και πληθωρισμού. Ξαναλέω, σε διάφορα κράτη-μέλη θα έχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Είναι λίγο πρόωρο να σας απαντήσω τώρα. Η επόμενη ερώτηση είναι της κυρίας Κέλλη. Μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο σημερίζεται την ανησυχία της, ε, ε, ε, του βουλευτή για το τελευταίο ευρωβαρόμετρο για τα μέτρα που χρειαζόμαστε για την καταπολέμηση της ανεργίας σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση χρειάζεται την νομιμοποίηση, χρειάζεται να ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με το τι κάνουμε. Εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερο βάρος στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση και στις δράσεις του. Θέλουμε να είναι αποτελεσματικές για την καταπολέμηση της ε, ανεργίας. Ε, και τα δύο εργαλεία είναι πάρα πολύ σημαντικά από οικονομική άποψη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ύφεση και να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση για την απασχόληση, να έχουμε μια καλύτερη στρατηγική και να αυξήσουμε τα προσόντα, ούτω ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι νέε θέσει ε, απασχόληση. Ε, το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήδη ανέλαβε ε, έκτατα μέτρα για την στήριξη τη απασχόληση. Το Συμβούλιο επιδιώκει η βελτίωση τη διαδικασία που θα ισχύει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ε, και έτσι ε, προτείνουμε να αναθεωρηθεί ο υφιστάμενος κανονισμός ε, για να υπάρχει αποτελεσματικότερη δράση για, τους, για όσους έπεσαν στην ανεργία λόγω της παγκοσμιοποίησης αλλά και λόγω της οικονομικής ύφεσης που όλοι βιώνουμε. Ε, επίσης να αναφέρουμε ότι για αυτό το ταμείο, πέρα από αυτό το ταμείο, χρειάζεται μια εκστρατεία ενημέρωσης ε, που είναι αρμοδιότητα και των κρατών μελών και της, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έκτε, Τα κράτη-μέλη πρέπει να ενημερώνουν για τις δράσεις, για τις συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ώστε να τονίσουν τον κοινοτικό ρόλο ε, και την υποστήριξη που προσφέρεται από τα ταμεία. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που, που δρομολόγησε σχετικά η Επιτροπή το 2005. Πρέπει να ε, υπάρχουν προσβάσιμες πληροφορίες ε, για όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ενημερώνονται όλοι οι δικαιούχοι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής ε, Συνοχής. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, επίσης θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν τους πολίτες τους και το ε, αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο θεσπίστηκε εσχάτως ε, και υπάρχει έλλειψη γνώσεων γενικά για αυτό το Ταμείο γιατί λίγες μόνο περιπτώσεις έχουν καλυφθεί από αυτό το Ταμείο το τελευταίο, τον τελευταίο χρόνο. Σας ευχαριστούμε. Ε, Ευχαριστώ για την πολύ σύντομη και πλήρη απάντησή σας. Θα ήθελα όμως να δευτερολογήσω. Αντιλαμβάνω ότι υπάρχει μεγάλη αντίθεση στο Συμβούλιο να χρηματοδοτηθεί το Ταμείο αυτό για τα επόμενα δύο χρόνια 100%. Το Συμβούλιο προτείνει κάποια εναλλακτική λύση για να διατηρήσουμε την όθηση προς τα εμπρός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του προγράμματος του θέματος. Ναι, είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως στο Συμβούλιο και υπάρχει ομόφωνη απόφαση ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα στοιχείο εθνικής χρηματοδότησης δηλαδή δεν πρόκειται το Συμβούλιο να στηρίξει την πλήρη χρηματοδότηση. Ζητήσαμε όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία εναλλακτική πρόταση και το συζήτησα προ δύο ημερών με τον υπεύθυνο επίτροπο και θα μας το υποβάλουν το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, η κυρία Τίκα έχει τον λόγο. με συγχωρείτε, αλλά στο Συμβούλιο δεν υπάρχει επαρκή στήριξη για να υποστηρίξουμε την καταπολέμηση της ανεργίας και να ε, χρηματοδοτηθεί 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Σε μία περίοδο κρίσεως, όταν ε, στα ναυπηγεία και στις χαλιβουργίες η ανεργία έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και ταχαίως είναι απαραίτητο να μπορέσει κανείς να εξασφαλίσει την ε, ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τι προβλέπετε για να μπορέσει το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Καταπολέμησης στην Παγκοσμιοποίηση ε, να στηρίξει ε, αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει εναλλακτικές προτάσεις όσον αφορά την χρήση αυτού του κοινωνικού ταμείου διότι όπως είπατε και εσείς υπάρχουν πολλοί άνεργοι στην Ευρώπη και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ταχαίως μία τέτοια πρόταση. Κάνουμε όμως και άλλα εναντίον της ανεργίας που είναι ευθύνη των κρατών μελών αλλά υπάρχει και συλλογική ευθύνη Προσπαθούμε να συντονίσουμε τις ενέργειες, να διευκολύνουμε την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, να καταργήσουμε τα εμπόδια, να μπορέσει από την 1η Ιανουαρίου να λειτουργήσει η οδηγία για τις υπηρεσίες και να δώσουμε ή στα άτομα που δεν μπορούν να βρουν δουλειά χρηματοδότηση να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους και να μπορέσουν να βρουν μια θέση εργασίας. Αυτά θα συζητηθούν στην άτυπη συνάντηση τον Οκτώβριο όπου η ανεργία είναι ένα από τα βασικά θέματα και ξέρω τέτοιες συζητήσεις γίνονται και στο Κοινοβούλιο και επηρεάζουν πολύ και την ε, μελλοντική εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι λοιπόν μόνο ένας τρόπος να ε, καταπολεμήσουμε ε, την ε, ε, ανεργία μεταξύ πολλών και θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα προχωράμε στο επόμενο ερώτημα του κυρίου Πόσελτ σχετικά με τις πληροφορίες για την Τσετσενία και το λόγο έχει υπουργό. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Μόλις ενημερώθηκε η Προεδρία για το φόνο της Νατάλια Εστεμίροβα Αμέσως ε, κάναμε μία δήλωση καταδικαστική και εκφράσαμε τα συλληπιτήριά μας για την οικογένειά της και για τους συναδέλφους της στην οργάνωση Memorial. Επίσης, ενημερώσαμε τις ρωσικές αρχές ότι πρέπει να κάνουν μία έρευνα για να επικρατήσει η αλήθεια και να επανορθωθεί η κατάσταση. Πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση στην Τσετσενία, κυρίως για την ε, κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Συμβούλιο επανειλημμένα ενθάρρυνα τις ρωσικές αρχές ε, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους ε, στην Ρωσία βάσει της σύμβασης του ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει παρουσία στην Τσετσενία. Στηρίζουμε προγράμματα και διπλωμάτες ε, από την ε, πρεσβεία μας ε, στη Μόσχα πηγαίνουμε τακτικά στην Τσετσενία και Φυσικά ανησυχούμε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία, αλλά δεν θεωρούμε ότι αιτιολογείται σήμερα να συσταθεί συγκεκριμένο γραφείο. Δεν υπάρχει εντολή ε, είμαστε παρόντες ε, στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση, να παρακολουθούμε συγγνώμη, την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών στην ε, Τσετσενία και κάθε φορά που χρειάζεται θα γύρουμε το ζήτημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Είναι η πρώτη καλή απάντηση που λαμβάνω από το Συμβούλιο επί του θέματος. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω συμπληρωματικά. Μπορεί το Συμβούλιο να ασχοληθεί συγκεκριμένο με, υπό την Σουηδική Προεδρία με την Τσετσενία συγκεκριμένα γιατί υπάρχουν ε, διάφορες ανακοινώσεις των ρωσικών αρχών ότι θα υπάρξουν αλλαγές τις οποίες ακούμε αλλά δεν βλέπουμε θα θέλαμε λοιπόν εφόσον πρόκειται να προετοιμαστεί η διαπραγματεύση για μια συμφωνία να υπάρξει αυτή η εξέταση και αύριο θα το αναφέρουμε και στα κατεπίκοντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα φιλικά σας λόγια, κύριε Πόσελτ. Ναι, ναι. Ε, διαρκώς, ε, ε, όταν έχουμε διάλογο με την Ρωσία, συζητάμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελπίζουμε το φθινόπωρο να γίνει σύνοδο κορυφή σε ΕΕ Ρωσία και φυσικά θα είναι στη μερίσια διάταξη το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση του κυρίου Χουντή ε, για την άδεια της ε, τουρκικής κυβέρνησης ε, για έρευνες υδρογονανθράκων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργέ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζει το Συμβούλιο τα τελευταία γεγονότα που υποδεικνύει ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή τους. Ε, σε αυτή την ε, περιοχή υπάρχει το θέμα των σχέσεων της Τουρκίας με άλλες χώρες ε, και φέρει ευθύνη και η Τουρκία για τις σχέσεις καλής γειτονίας. Έτσι προβλέπεται και από τον ΟΗΕ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προσχώρηση της Τουρκίας. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και στα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία να αποφύγει να δημιουργεί συγκρούσεις και να κάνει πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας ε, και τη διαδικασία ειρηνική επίλυση των διαφορών. Επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι πρέπει να ε, ομαλοποιηθούν οι διμερεί σχέσει τη Τουρκία με όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένε και τη Κύπρου και όλα φυσικά τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά για το ίδιο. Ε, Προ το πρωτόκολλο γνωρίζετε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεφέρει ευθύνη η Τουρκία για την πλήρη υλοποίηση του πρωτοκόλλου χωρί καμία διάκριση. Ε, και συστηματικά αναφέρεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί διευθυντέ ε, που συναντήθηκαν στο Χόλμη το Ιούλιο το συζήτησαν και στο Συμβούλιο Σύνδεση ε, στο Μάιο συζητήθηκε το θέμα. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τι εξελίξει. Παρακαλώ, κύριε <clears throat> Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ εκτιμώ και τη διάθεσή σας και το κουράγιο σας να δώσετε σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε. Ε, θέλω να σας πω ότι αύριο το Κοινοβούλιο θα συζητήσει το θέμα του αγωγού του Ναμπούκο αφού σας θυμίσω ότι τον Ιανουάριο του 2009 ο Τούρκος Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες είχε απειλήσει ότι η χώρα του θα επανεξετάσει τη στήριξή της στην κατασκευή του, του αγωγού φυσικού αερίου αν δεν συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το άνοιγμα του κεφαλαίου ενέργεια αυτό το κεφάλαιο όπως ξέρετε έχει μπλοκαριστεί από το βέτο που έχει ασκήσει η κύπρος επειδή έχει απειληθεί από την τουρκία για την εκμετάλλευση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. επειδή λοιπόν το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι κρίσιμης σημασίας και ενδεχομένως δημιουργήσει μείζωνα προβλήματα σε πολλές πολιτικές της ευρωπαϊκής ένωσης σας ερωτώ και πάλι κυρία υπουργέ τι μέτρα θα λάβει το συμβούλιο για να αναγνωρίσει η τουρκία το δικαίωμα στην κύπρο σε αποκλειστική οικονομική ζώνη. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνουν όλες τις παρατηρήσεις και ξαναλέω θα παρακολουθήσουμε ε, τις εξελίξεις ε, και φυσικά σε όποιες επαφές έχουμε ε, με την Τουρκία θα τονίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι καλές σχέσεις γειτονίας. Έχουμε και την Τρόικα τον Νοέμβριο και ελπίζω ότι τέτοια περιστατικά θα μπορέσουν να αποφευθούν στο μέλλον. Για το κεφάλαιο ενέργεια τώρα για τις διαπραγματεύσεις, Συζητείται το θέμα σε διάφορε συνθέσει του Συμβουλίου. Είναι λίγο πρόωρο ε, να προδικάσουμε το αποτέλεσμα τη αξιολόγηση τώρα και όπω γνωρίζει ο αξιότιμο βουλευτή, κάθε βήμα σε αυτή τη διαδικασία ε, απαιτεί την ε, ομοθυμία στο Συμβούλιο. Next question, Περνάμε στο επόμενο, στην επόμενη ερώτηση. στην ε, ε, ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βερμανία. Ευχαριστώ να βρω το σωστό χαρτί. Παρακολουθούμε ε, προσεκτικά την κατάσταση από τότε που τη φυλακίσαν την Αung Σουική πριν από 20 χρόνια και ε, συνεχώς ε, ενθαρρύναμε τις βυρμανικές αρχές να την απελευθερώσουν τότε εγκρίναμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Θα παριθμίσω κάποια από αυτά. Τον Αύγουστο ε, καταδικάσαμε την απόφαση κατά της Aung San Suu ε, γιατί δεν υπήρχε νομική βάση για την ε, καταδίκη της και ενθαρρύναμε τις βιρμανικές αρχές να την απελευθερώσουν χωρίς κανέναν όρο και αναφέραμε ότι συνιστά η καταδίκη της παραβίας του εθνικού και του διεθνούς δικαίου. Ο Ξαβιέ Σολάνα, τους εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην Σύνοδο Κορυφής ε, του ΑΣΕΑΝ, ε, αναφέρθηκε στο θέμα και επίσης τον Ιούλιο στη Σύνοδο Κορυφής ΑΣΕΑΝ Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκε το θέμα παρουσία του εκπροσώπου της Βυρμανίας. Σε αυτή τη σύνοδο αναφέρθηκε ισχυρή απέτηση όλων των ΗΠΑ ε, της ε, Κίνας, ε, της Ρωσίας να απελευθερωθούν πάρα αυτά όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Επίσης δραστηριοποιούμαστε με τον κύριο Φασίνο, τον ειδικό επισταλμένο μας στην Βιρμανία και έχουμε και τον ειδικό σύμβουλο, τον Ιμπρέμ Καμπάρη του ΟΗΕ που έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και με, συνεργαζόμαστε και με άλλους εταίρους στην Ασία αλλά όλες οι διαμαρτυρίες αγνοήθηκαν από τις Βυρμανικές αρχές παρότι ε, υπευλήθησαν ε, αιτήματα από διάφορε χώρε από διάφορου ε, διεθνού οργανισμού, από τον πρόεδρο του ΑΣΕΑΝ, από τον ΟΗΕ, από διάφορα κράτη-μέλη του ΑΣΕΑΝ και μην ξεχνάτε ότι η Βυρμανία ανήκει στον ΑΣΕΑΝ. δεν υπήρξε απάντηση λοιπόν από τις βυρμανικέ αρχές και εμείς αναλάβαμε μέτρα κατά των υπευθύνων καταδικάσαμε μέλη του δικαστικού σώματος και άλλων που εμπλέκονται στην υπόθεση της ε, Aung San Suu Kyi ε, και ε, διατάξαμε πάγωμα των περιουσιακών τους ε, στοιχείων ε, και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε περιοριστικά μέτρα ε, και με πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων που υποστηρίζουν το καθεστώς στη Βυρμανία και όλων των σχετιζόμενων ατόμων. Και εκφράσαμε τη θέση μας στις 30 Αυγούστου που συνάδει πλήρω με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου από πέρσι. Σας καθησυχάζω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από όλα αυτά τα πολύ ειδικά μέτρα θα εντυπωποιήσει ε, τη συνεργασία της ε, με τη διεθνή κοινότητα, ε, κυρίως με τους ομοτήμους μας στην Ασία, ούτως ώστε πάρα αυτά να απελευθερωθεί χωρίς κανέναν όρο όχι μόνο η Αουν αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί ε, κρατούμενοι. Ε, χρειάζεται διεθνής ε, συντονισμός, αλλιώς δεν θα είναι ε, ισότιμες και αξιόπιστες οι εκλογές που θα γίνουν το 2010. Ευχαριστώ, κύριε ε, Πρόεδρε, για την εκτενή απάντηση. Παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε τι προσπάθεια γίνεται για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν προς την ε, Κίνα λόγω της διαμάχης μεταξύ της Χούντας και των εθνικών μειονοτήτων. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Θα επανέλθω επί του θέματος, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Και τώρα προχωράμε στο επόμενο ερώτημα του κυρίου Κρόλη σχετικά με τις χενότερες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ηνωμένων Πολιτειών. Η Υπουργός. Eh, eh. Ευχαριστούμε κύριε Κράουλη. Ε, το Συμβουλίο αποδίδει ιδιαίτερο βάρος ε, στις σχέσεις ΕΕ, οι διατλαντικές σχέσεις. Είναι ακρογωνίως λίθος εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε κοινές αξίες, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και δέσμευση για ε, ανοιχτές και ολοκληρωμένες οικονομίες. με τη νέα κυβέρνηση στη ΣΥΠΑ τονώθηκαν οι σχέσεις και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία ε, γιατί τώρα περιμένουμε αυτά αποτελέσματα της διατλαντικής ε, σχέσης ε, αφωτέρων των πλευρών και υπάρχουν πολλοί τομείς όπου συνεργαζόμαστε στενά με τη ΣΥΠΑ για να διευρύνουμε τις στρατηγικές εταιρικέ μας σχέσεις και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία σε διάφορα περιφερειακά ζητήματα Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράν ε, ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Ρωσία, ε, ε, Δυτικά Βαλκάνια, διαχείριση των κρίσεων και σε αυτόν τον τομέα συνεργαζόμαστε και χαιρόμαστε που συμμετέχουν οι ΙΠΑ στο, στην, στους που έχουν στείλει στο Κωσυφοπέδιο που έχουν σταλεί από τον ΟΗΕ στο Κωσυφοπέδιο και με τη νέα κυβέρνηση Ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και στον τομέα του περιβάλλοντο, ε, κυρίω το πρωτόκολλο του Κιώτο και την μείωση των εκπομπών ε, των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Για τα ενεργειακά ζητήματα θεωρούμε ότι πρέπει να ανέβουν σε ανώτερο επίπεδο, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ειδικό ενεργειακό συμβούλιο, ΕΕ, είπα, ένα ειδικό φόρουμ για να συνεργαστούμε για την ενεργειακή ασφάλεια, τι ενεργειακέ αγορέ, την πολιτική τη βιωσιμότητα και την έρευνα για τι νέε τεχνολογίε και νέε πολιτικέ άλλο ζήτημα φυσικά. Η χρηματοπιστωτική κρίση εδώ χρειάζεται στενή συνεργασία, ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη που έχουν οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ και να αποκαταστήσουμε την εύρυθμη λειτουργία του. Ε, έχουμε και το γύρο τη Ντόχα. Ε, πρέπει να περατωθεί το 2010 επιτυχώ. Είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάκαμψη και για την καταπολέμηση του προστατευτισμού ε, και φυσικά είναι σημαντικό εταίρο μα, είπα, σε αυτό το τομέα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 Ε, θα συζητηθούν φυσικά την ερχόμενη εβδομάδα στην, ε, τα συζητήματα αυτά στη σύσκεψη του G20 και ε, είναι προς κοινό μας συμφέρον να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας και να κατανοήσουμε το νομικό πλαίσιο και το κεκτημένο ημέν των δε. Μην ξεχνάτε τη φυλακή του Αγκαντανόμου τη συνεργασία μας στην, στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Έχουν, έχει ήδη γίνει ένα σημαντικό βήμα. Ε, επίσης είναι σημαντική συνεργασία για τον αφοπλισμό και ε, βλέπετε την αλλαγή της τάσης σε σχέση με την Κούβα ε, και ε, έχουν γίνει σημαντικά ζητήματα για την σύμβαση για τη μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και ε, έτσι ε, μπορεί να αποτελματωθεί ε, η κατάσταση στη σχετική διάσκεψη και να συζητηθούν και τα θέματα των πυρηνικών υλικών που χρησιμοποιούνται από τους ΜΕΝ και τους ΔΕ. Πρέπει να ενισχύσουμε τον διατλαντικό διάλογο να αυξήσουμε τη συνεργασία μας. Ε, έχουμε κοινό συμφέρον ε, να ε, βελτιώσουμε τις δράσεις μας στον αναπτυξιακό τομέα και στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ θα έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και άλλα συναφή σε ανώτατο επίπεδο και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που ε, θα ε, ηγηθούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την σύνοδο. Είμαστε πεπισμένοι ε, ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έναν λίγο επικοδομητικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ κύριο Σκρόλη. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ Σεσίλια. Με τα χαρά σας ξαναβλέπω εδώ με διαφορετικό καπέλο. Ε, μπορούμε καταρχήν να συνεργαστούμε ε, ενάντια τη, υπέρ του αφοπλισμού ε, και στις οικονομικές σχέσεις διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν συγκεκριμένες ιδέες για τα θέματα τα οποία θα φέρουν εις το επικείμενο συμβούλιο το οποίο πρόκειται να οργανωθεί μεταξύ των δύο αυτών ενωτήτων και ε, θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας τις γαλλικές ιδέες και τις αγγλικές ιδέες που παρουσίασε χθες ο Gordon Μπράουν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα το πρωί έγινε μια συζήτηση για την προετοιμασία του G20 και ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν διάφορες προτάσεις που έχουν συζητηθεί στον τύπο αλλά είμαστε καλά συντονισμένοι, έχουμε συζητήσει με τους υπουργού Οικονομικών αύριο το βράδυ θα έχουμε ένα γεύμα με τους Πρωθυπουργού και αρχηγούς κρατών για να καταλήξουμε στις θέσεις μας εν του Πίτσμπεργκ. Θα υπάρξουν προτάσεις αποφάσεις υπάρχουν ήδη και θα γίνει και ο τελικός συντονισμός αύριο. Δεν ανησυχώ γι' αυτό και ελπίζουμε ότι με την βοήθεια της Επιτροπής και του Επιτρόπου Αλμούνια έχουμε επιτύχει αυτό το σπάνιο επίτευγμα ομοφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συζητήσουμε τις πρωτοβουλίε μας και ε, τις ε, ιδέες μας μαζί με την Αμερικανική Διοίκηση και τους άλλους που θα συμμετέχουν στην συνάντηση των G20 για την μη επέκταση των πυρηνικών εξοπλισμών είναι το κατάλληλο σημείο να συζητηθεί και χαιρόμαστε για την προσήλωση δήλωση του Πρόεδρου Ομπάμα επί του θέματος αλλά θα χρειαστεί ε, χρόνο υπάρχουν ε, περίπλοκες ε, περίπλοκα θέματα τα οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε δεν ξέρουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί ε, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμά μας ελπίζουμε ότι θα τα προωθήσουμε και ε, ελπίζουμε ότι θα μας προσεγγίσουν και οι Αμερικάνοι σε αυτό. Ευχαριστώ. Μία ακόμη επιπρόσθετη ερώτηση από τον κύριο Παλέκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά το τρίγωνο Ευρωπαϊκής Ενώσεως είπα και Ρωσίας διότι Ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει ε, σοβαρές διαπραγματεύσεις ε, για τον πυρονικό αφεπλισμό πώς μπορεί να διευκολύνει η Ευρώπη και να επηρεάσει αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και τις διαπραγματεύσεις που έχουν μεγάλες επιπτώσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Λοιπόν, Είμαι πολύ ευτυχής για αυτά τα νέα. Είναι πολύ βασικό αυτές οι δύο χώρες να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα βασικά θέματα για την ανθρωπότητα και να προχωρήσουν. Βεβαίως υπάρχει μία διάσκεψη κορυφής ε, για τα πυρηνικά θέματα το Μάρτιο του 2010 όπου θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η κατάλληλη στιγμή να συντονίσουμε τις ιδέες μας και να δούμε πώς μπορούμε εμείς να, επιτυχ... να συμβάλλουμε στην επιτυχία αυτών των συζητήσεων. Ευχαριστώ. Προβλέπετε ότι θα τελειώσει ο χρόνος των ερωτήσεων στις 7 και η υπουργό πρέπει να φύγει. Όσες απαντήσεις δεν δόθησαν θα δοθούν γραπτώσεις στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Λίγη ο χρόνος για η ε, συνεδρίαση και η επόμενη συνεδρίαση θα ξεκινήσει αύριο το πρωί στις 9 ε, μέχρι τη 1 και 3 ε, με 7. Υπάρχει